witam panów posłów. επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. καλώς ορίσατε. όλοι οι παρόντες και εσείς κύριε επίτροπε καλώς ορίσατε. τα χτεσινά συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν διατίθενται. Έχετε σχόλια, παρατηρήσεις για τα συνοπτικά πρακτικά. Όχι.